πια από τα προγράμματά μας και θα έχει επικρατήσει και καθεστώς απελευθερωμένο όσον αφορά τις θεωρίες διαβατηρίων. Αλλά η Ουκρανία πρέπει να κάνει τις μεταρρυθμίσεις. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κολάρσκα. Περνάμε τώρα στην οφθαλμοθυρευτική διαδικασία. Ο κύριος Σφόμποντα έχει ήδη κάνει πολλές τέτοιες παρεμβάσεις αυτού του είδους. Είναι ίσως λιγότερες παρεμβάσεις από ό,τι φοβόμαστε στην αρχή, αλλά περισσότερες από ό,τι μπορούμε να αποδεχτούμε. Δίνω λοιπόν τον λόγο στον κύριο Κοσλόφσκι πρώτα. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι.